νομικές πράξεις, οι τίτλοι των οποίων επίσης θα δημοσιευτούν στα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης. Περνάμε τώρα στην έγκριση της ημερήσιας διάταξης για αυτή τη...